Έχετε το λόγο. Λυπάμαι πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπαινοβγαίνει κόσμος στην αίθουσα. Υπάρχουν πολλές κουβέντες σαν να είναι καφενείο. Αυτό είναι προσβολή κατά των ψηφοφόρων, κατά των πολιτών που πρέπει να κάνουμε ομιλίες σε αυτό το περιβάλλον. Παρακαλώ να εξασφαλίσετε ότι επικρατήσει ηρεμία και ησυχία και μετά μπορούμε να μιλήσουμε. Και δεν ξέρω για ποια επεξήγηση ψήφου μιλάμε, διότι ο πίνακας δεν δείχνει. Σας παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη να μπορούμε να βλέπουμε τι συμβαίνει και να μπορούμε και να ακουγόμαστε, διότι σε αυτή τη φάση δεν ακούω τίποτα και δεν βλέπω και τίποτα. Και σαν Πρόεδρος παρακαλώ να εξασφαλίσετε ότι όλα είναι όπως πρέπει. Κυρία Μορβάη, λοιπόν, λυπάμαι. Για τεχνικούς λόγους υπήρχε το πρόβλημα. Τώρα μιλάμε για την έκθεση Becker. Και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την έκθεση αυτή. Πρόκειται λοιπόν για την ε, περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς εργασίας και για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν κινητικότητα στους εργαζομένους. Όταν πρωτοείδε αυτή την έκθεση θεώρησα ότι είναι θαυμάσιο το ότι θα ενοποιηθούν επιτέλους οι αγορές εργασίας, επιτέλους οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Άγγλοι γιατροί και νοσοκόμες θα έρθουν στην Ουγγαρία. Κατά ε, ορδές θα έρθουν και θα λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ουγγαρία για την περίθαλψη θα μπορέσουμε να φροντίσουμε τους ασθενείς μας όπως ε, χρειάζεται. Θεωρούσα λοιπόν ότι επιτέλους πολλοί άλλοι οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα έρθουν από τη Δυτική Ευρώπη προς την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι δεν θα είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ε, αποκαλούμε αυτή την κατάσταση ενοποίηση των αγορών εργασίας, γιατί η κινητικότητα είναι ε, μόνο προς ε, τα μία κατεύθυνση, άρα είναι φυγή εγκεφάλου. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ πολύ. Η πολιτική απασχόληση είναι πολύ σημαντικό τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ο εξορθολογισμός της κινητικότητας και η ενοποίηση της αγοράς εργασίας είναι κάτι το πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ε, όταν ε, εργάζονται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα να έχουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και ανεξάρτητα ε, από την υπηκότητά τους. Οπότε δεν θα πρέπει να προκύψει καμία διάκριση και χαιρετίζω το ότι ε, το έχετε βάλει αυτό στην έκθεση. Πρέπει να ε, ε, καταλάβετε ότι πολλοί έχουν λάβει βοήθεια και ότι πολλοί εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν βοήθεια και πιστεύω ότι χρειάζονται πολλές περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Σογκόρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για την ενίσχυση της κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να επιτύχουμε περισσότερη απασχόληση. Εγώ θεωρώ ότι η στόχη αυτή είναι πολύ σημαντική, αλλά θέλω επιπλέον να προσθέσω ότι αυτό πρέπει να πάει παράλληλα με την ενίσχυση της ε, συνοχής μέσω πιο αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής και ότι τα ανατολικά κράτη-μέλη πρέπει να καλύψουν την καθυστέρησή τους. Αυτή τη στιγμή από την ε, ανατολική περιφέρεια της Ένωσης πηγαίνουν ε, στην ε, Δυτική και δεν πηγαίνουν εκεί για να πάρουν επιδόματα γιατί μπορούν να κερδίσουν περισσότερα. Στη Ρουμανία οι δάσκαλοι παίρνουν 300 ευρώ το μήνα παρά το ότι οι υπηρεσίες και πολλά προϊόντα έχουν την ίδια τιμή όπως και στη Δύση. Λόγω αυτών των περιστάσεων δεν μπορούμε να αποκαλέσουμε αυτή τη διαδικασία ενοποίηση της αγοράς εργασίας και όχι δεν μπορούμε να την αποκαλέσουμε ευρωπαϊκή αγορά εργασία. Αν δεν καλύψουν την καθυστέρηση τα φτωχότερα κράτη-μέλη, θα υπάρξουν μεγαλύτερα κύματα μετανάστευση. Οπότε θα αυξηθούν τα χάσματα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σάρνοτ, στο Ηνωμένο Βασίλειο το θέμα της μετανάστευσης και η κρίση των προσφύγων ε, ε, ε, λοιπόν, έρχονται μετανάστες και όχι οι πρόσφυγες. 96% είναι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλούς ανειδίκευτους στον Ηνωμένο Βασίλειο και η Τράπεζα της Αγγλίας που λέει για 10% σε μετανάστευση σε κάποιους τομείς περικόπτονται κατά 1,8% οι αμοιβέ. Και στα βορειοδυτικά της Αγγλίας, στην περιοχή, μόνο ακόμα χειρότερα. Έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία στη χώρα. Λοιπόν, η σημερινή ψηφοφορία για τα κέντρα απασχόλησης που θα πρέπει να διαφανίζουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κενέ θέσει για βιογραφικά που ταιριάζουν κλπ. θα οδηγήσει περισσότερο να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βεβαίω ο κόσμο ήδη πηγαίνει, διότι τα αγγλικά είναι και παγκόσμια γλώσσα. Μπορεί να ξεχάσουμε την κατεπίγουσα ανάγκη. Διότι με μία ψηφοφορία κάναμε τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά και παρόλα αυτά φαίνεται τελικά και το εργατικό κόμμα αισθάνεται άνετα να ψηφίσει αυτά τα μέτρα. Μετά έχουμε επεξήγηση ψήφου, λέει Πρόεδρος, που αφορά την εισαγωγή μέτρων κατεπηγόντων αυτονόμων για την, νησία. Και η πρώτη που θα πάρει το λόγο είναι η κυρία Μπεσέρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την Ισία έχει πραγματοποιήσει σημαντική δημοκρατική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και είναι κύριο εταίρο Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπαγκρέπ. Παράδειγμα ε, επιτυχίε τη Αραβική Άνοιξη. Θα πρέπει να στηρίξουμε την Τινησία σε αυτή την προσπάθεια υπέρβαση που κάνει. Γι' αυτό και τάχθηκα και υπερψήφισα αυτά τα μέτρα τα αυτόνομα. Αλλά δεν συμφωνώ με τι τροπολογίε που υιοθετούν μια πιο προστατευτική στάση για το ελαιόλαδο. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, Ισπανικής Καταγωγής φυσικά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κάνουμε μια αξιολόγηση του αντικτύπου των μέτρων αυτού του ψηφίσματο ό,τι αφορά τον προστατευτικό χαρακτήρα για το ελαιόλαδο και φυσικά να δούμε ε, πώς θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της Τινησίας. Ε, κρίμα που δεν υπάρχει μια μόνιμη μία του γεγονότος ε, της, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τινησία στο ε, ανώτατο επίπεδο και να σταματήσουν οι παρενοχλήσεις προς την κοινότητα ομοφιλοφίλων ε, ε ΛΟΑΔΜ γενικώ. Γιατί αυτό είναι μία μάστιγα και θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η παρενόχληση. Η κυρία Σένερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή γιατί είμαι βεβαία ότι τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να βοηθήσουν ούτε το λαό ούτε τους γεωργούς της Τινησίας. Αλλά απλώς είναι μέτρα για να γίνει πιο φθηνή η ελιά, κάτι που θα πλήξει τους μικρομεσαίους παραγωγούς και των χωρών του Νότου αλλά και, των, και της Τινησίας. Επίσης ε, δεν δίνεται κανένα εχέγγυο ότι το ελαιόλαδο της Τινησίας δεν θα, διατεθεί, δεν θα διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά με τιμή κάτω του κόστου σε οικονομικό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από τότε που πριν από πέντε χρόνια άλλαξε το καθεστώς στην Τινησία, ε, εισήχθησαν μακροπρόθεσμες ε, μεταρρυθμίσεις και υπάρχει αναδιάρθρωση της κοινωνίας. Αλλά κάποιοι τομείς που είναι πολύ σημαντικοί και εξακολουθούν να είναι βασικοί για την οικονομία της χώρας, όπως είναι η παραγωγή ελαιολάδου. Πριν από την ε, Επανάσταση, η Τινησία ήταν ο έβδομος παγκόσμια μεγαλύτερος παραγωγός όμως σήμερα αποφασίσαμε να στηρίξουμε τη Ισία Είναι ένα σύστημα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξη 35.000 τόνοι το χρόνο για δύο χρόνια μέχρι το 17 και αυτό γιατί είναι σημαντικό εταίρο μας στην Ισία και με τα μέτρα αυτά θα προωθήσουμε τη σταθερότητα και την εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόλτσακ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα επίσης την έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι σίγουρα θα πρέπει να εκτιμήσουμε την πρόοδο που έχει πετύχει σε πέντε χρόνια η Τινησία ανήκει στη λέσχη των δημοκρατικών κρατών η χώρα τώρα αυτή πρέπει να εκτιμήσουμε την πρόοδο της χώρας και αυτή η εικόνα θα πρέπει να επικρατήσει έναντι των συνεπειών που έχουν τα μέτρα αυτά για κάποιους παραγωγούς ελαιολάδου Απ' την άλλη θα πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα αυτή καθεαυτή παρά το ότι αυτή η πράξη έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες λόγω της αύξησης του ελευθέρου εμπορίου. Αλλά νομίζω ότι είναι το τίμημα αποδεκτό αν θέλουμε να βοηθήσουμε την Τινησία. Κύριε Κέλλη, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό το σημείο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψήφισα με την ομάδα με αυτή την έκθεση. όπως έκαναν και άλλοι ε, και 123 ψήφισαν κατά της εκθέσεως. Είναι σημαντική έκθεση, πρέπει να δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια στην Τινησία. Και χρειάζονται αυτά τα κατεπήγοντα μέτρα τα εμπορικά για την Ισία... Είναι κάτι πολύ σημαντικό και κρίσιμο σε αυτή τη φάση, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής ε, θέσεως της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε έναν κανονισμό που προσφέρει μονομερές ε, άρσεις δασμών για τις εξαγωγές τη. Ε, για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτονόμων εμπορικών μέτρων. Αυτό έχει νόημα ε, και ένα εκατομμύριο άνθρωποι έμεσα ή άμεσα ανα, ε, αναμειγνύονται στην παραγωγή του ελαιολέδου και θα πρέπει να γίνει διάμεση αξιολόγηση συνεπιών να δούμε πώς τα μέτρα αυτά επηρεάζουν και τους δικούς μας παραγωγούς ελαιολάδου στην Ευρώπη και αν έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, αρνητικό αντίκτυπο ίσως θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε διορθωτικά μέτρα. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο σημείο. Έκθεση Μαρία Ζωάου Ροντρίγκε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για Οικονομική Πολιτική. Η κυρία Μορβάη είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Έχει το λόγο, κυρία Μορβάη. Κοιτάξτε, ελάχιστε αλλαγέ έχουμε όσον αφορά τον ήχο στην αίθουσα, την έλλειψη ησυχία. Είμαι ένα από αυτού που δεν μπορώ να μου παράλληλα όταν μιλάνε κι άλλοι δυνατά. Για μία ακόμη φορά σας παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη να ζητήσετε σε εκείνους που θέλουν να συνομιλούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα και να αφήσουν τους άλλους που θέλουν να κάνουν ομιλίες ε, να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις ομιλίες. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τη δική μου γλώσσα. Λοιπόν, θέλουμε να αποτιμήσουμε την ε, οικονομική ανάπτυξη για το 2016. Σε σχέση με αυτό, θέλω να πω ότι δεν υπερψήφισα την έκθεση και παρακαλώ την Αντιπρόεδρο αυτό να μην ε, υπολογιστεί στο χρόνο ομιλίας μου. Να μην σταματήσει δηλαδή τώρα η ομιλία μου. Ε, στην Ουγγαρία μία οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν ακόμη να λειτουργήσουν όπως μου είπε ένας επικεφαλής μιας οικογενειακής επιχείρησης και μπορεί να ζήσει στην κοινωνία του. Επίσης μου εξήγησε ότι ελπίζει και τα εγγόνια του να μπορέσουν μια μέρα να αναλάβουν την επιχείρηση και ότι η επιχείρηση δεν θα χρειαστεί και ότι τα εγγόνια του αυτά δεν θα χρειαστεί κάποια στιγμή λοιπόν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να βρουν δουλειά. Αυτό είναι το μέλλον για τη χώρα μας και όχι αυτή η οικονομική ανάπτυξη όπως τη περιγράφετε εσείς. Δεν πιστεύω σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ο κ. Γκονζάλης ο Ο κ. Μάμικινς και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πυλώνας ε, για την επιβίωση της Ένωσης και γι' αυτό αυτή η έκθεση για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να υποστηριχθεί. Χρειάζεται ανταλλαγή απόψεων, οικονομικές μεταρρυθμίσεις και πολλές άλλες πλευρές για να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά θα μας ωφελήσουν όλους και με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε την οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι οι επενδύσεις, η φορολογική πολιτική και οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμπληρωθούν με αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. Ε, η ελεύθερη αγορά είναι αυτονόητη. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η ζήτηση έχει ειδικά χαρακτηριστικά γιατί παίζουν ρόλο σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ. Και πάλι ψήφισα όπως και η υπόλοιπη ομάδα μου και ξέρω ότι ήταν μεγάλη πλειοψηφία, τα δύο τρίτα συγκεκριμένα που υπερψήφισαν και ένα τρίτο που καταψήφισε. Χαίρομαι για τις φιλόδοξες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν και κυρίως για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την ενίσχυση της οικονομικής ε, σύγκλησης με την ενίσχυση και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ε, ε, για παράδειγμα, η παράγραφος 16 μιλά για την νεόθεση στις επενδύσεις, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό των οικονομιών και φυσικά μιλά για υπεύθυνε και όχι λαϊκιστικές και δημαγωγικές δημοσιονομικές πολιτικές. Επίσης, χαίρομαι για τη δέσμευση να μειωθεί η μακροχρόνια ανεργία και ιδιαίτερα τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων. Αν καταφέρουμε να ελοπίσουμε όλους αυτούς τους στόχους, πραγματικά θα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Ο κύριος Σουλίκ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ďakujem Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς ε, καταψήφισα αυτή την έκθεση. Επικρίνεται η μαύρη αγορά εργασίας σε αυτή την έκθεση και ε, προτείνονται βήματα που θα κάνουν την νόμιμη απασχόληση πιο ακριβή. Χρειαζόμαστε πραγματική ανάπτυξη και ανακατανομή του πλούτου επικρίνεται υπερχρέωση και προτείνονται πολλά μέτρα τα οποία θα αυξήσουν την υπερχρέωση. Η έκθεση λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει τρομερή ανεργία, αλλά παράλληλα αυξάνεται η ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή και αυτό θα αυξήσει περισσότερο την ανεργία. Μπορούμε να γράφουμε συνέχεια εκθέσεις αλλά η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερη ελευθερία, λιγότερη ανακατανομή. Ένα λεπτό, κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους. Για πραγματικούς ανθρώπους αποφασίζουμε που ζουν στις χώρες μας. Και επανέρχομαι και στην ιστορία που σας είπα για μια οικογενειακή επιχείρηση μίλησα με κάποιον που εργάζεται σε μια οικογενειακή επιχείρηση και όχι σε πολυεθνική. Και αυτός ο επιχειρηματίας μου είπε ότι θέλει να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται και να διατηρηθεί η οικογενειακή του επιχείρηση. Θέλουμε να την υποστηρίξουμε λοιπόν και εμείς αυτή την επιχείρηση. Αυτή η δεύτερη έκθεση ασχολείται με κοινωνικά μέτρα και μέτρα αύξησης της απασχόλησης. Όμως εάν εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση άνθρωποι πολλά προβλήματα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ανεργία για παράδειγμα. Διότι η οικογένεια θα κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε όλα τις τα μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται. Δεν πρόκειται κανένας να ε, ε ρίξει κάποιον στον δρόμο από την οικογένειά του. Είτε είναι νέες μητέρες, είτε είναι γυρεότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πρέπει να υποστηρίξουμε τη στεγαστική πολιτική και πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την ανακαίνιση των κατοικιών, για την περίθαλψη, για τους νέους, για τους ηλικιωμένους. Να διάφοροι τομείς. Όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να ενισχυθούν. Είναι απόλυτα αναγκαίο για ολόκληρη την Ένωση και φυσικά και για τη χώρα μου, τη Λετωνία. Και ιδίω πρέπει να αναφερθώ στην πολιτική για τους νέους και τα παιδιά. Διότι αν δεν φροντίσουμε για το σπίτι μας, για τον κήπο μας, αν δεν φροντίσουμε τη σωδιά μας, δεν θα έχουμε αρκετά τρόφιμα. Μόνο έτσι θα αποδώσει η εργασία μας. Τα παιδιά είναι το πιο όμορφο που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να τα καλλιεργήσουμε και αυτά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, για να έχουν ένα μέλλον. Γι' αυτό υποστήριξα αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όγκορ. Κοιτάξτε, έχουμε μικρή ανάπτυξη και μειώνονται κάπω η ανεργία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ κρατών μελών και υπάρχουν διαθετικά προβλήματα όσον αφορά την αγορά εργασία. Το ποσοστό οικονομική ε, ανάκαμψη χαμηλότερο από αυτό που θέλουμε. 20% είναι η ανεργία των νέων. Η μακρά διαρκεία ανεργία που έχει διπλασιαστεί είναι ανησυχητική. Δημιουργείται σοβαρό κίνδυνο έτσι για φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στι κοινωνίε μα. Ε, και επιδεινώνεται η κατάσταση αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Γι' αυτό καλωσορίζω την έκθεση που ζητά πιο υπεύθυνε διαθετικέ μεταρρυθμίσει και περισσότερε επενδύσει για το ανθρώπινο κεφάλαιο, τους, ώστε να αναπτυχθεί ανθεκτική οικονομία και αγορά εργασία που συμβαίνει του πάντε και να μπορεί να αντέχει στι προκλήσει λόγω τη αυξήσεω του πληθυσμού και λόγω τη ε, μεγαλύτερη οικονομική εξάρτηση που δημιουργείται. Ευχαριστώ. Τελευταίο για αυτό το θέμα ο κύριο Μάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όποιος ε, θεωρεί ότι δεν έχει μέλλον η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ένωσης, έχει λάθος. Διότι θα έχουμε 2% αύξηση φέτος. Η ανεργία επιτέλους θα μειωθεί. Τα πολιτικά μέτρα που λάβαμε σιγά σιγά έχουν επίδραση. Τα μέτρα για τους νέους, οι εγγυήσει και το πρόγραμμα απασχόλησης εφαρμόζονται με συνέπεια και τα κράτη-μέλη επιτέλους καλύπτουν τις καθυστερήσεις τους. 4,8 εκατομμύρια νέοι που ψάχνουν για μαθητεία ή για δουλειά δεν θα πρέπει να αφαιθούν στην τύχη τους. Η έκθεση Ριμπέρο αναφέρεται και σε συγκεκριμένου δείκτε που πρέπει να έχουν το ίδιο καθεστώ όπω και οι οικονομικοί δείκτε. Είναι κοινωνικοί δείκτε. Πρέπει λοιπόν να συνοδευτούν από βαθιέ αναλύσει για τα συγκεκριμένα προβλήματα στι διάφορε χώρε μέλη. Εάν δράσουμε αποτελεσματικά, θα καταπολεμήσουμε και την ανεργία και την απόγνωση και τον αποκλεισμό. Έτσι θα δείξουμε τις αξίες μας, αλληλεγγύη, ανθρωπισμό στις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Έκθεση της κυρίας Καθρίν ε, Στάιλερ για τη διακυβέρνηση στην ενιαία αγορά εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η κυρία Μορβά είναι η πρώτη μας ομιλήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να φτιάξω ένα λεξικό που να περιέχει ε, ε, το λεξιλόγιο για την ε, Ανατολική Ευρώπη της Ένωσης. Τι σημαίνει ενιαία αγορά για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Για μας σημαίνει ότι είμαστε ανοιχτοί για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, ότι πρέπει να τους δώσουμε όλες μας τις επιχειρήσεις, ότι πρέπει να τους δώσουμε όλη μας τη γη ότι στους Γάλλους και στους Γερμανούς πρέπει να τους δίνουμε τα πάντα. Κάθε δυνατότητα που έχουν οι χώρες μας. Να είναι ανοιχτές όλες μας οι επιχειρήσεις για αυτούς. Και οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι θέλουν για αυτούς. Και δεν μπορούμε να ε, ευνοήσουμε τους δικούς μας ε, ενιαία αγορά. Σημαίνει και οι ουγγρικές επιχειρήσεις να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως και οι δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Ουγγαρία. Πιστεύω ότι πρέπει να πούμε τα πράγματα του όνομά του και εδώ πρόκειται για πικιοκρατία. Ευχαριστώ. Τι είναι σημαντικό, λέει ο κύριος Μαμίκιν σε αυτή την έκθεση. Πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα συστήματα τυποποίησης πρέπει να ανακαινιστούν. Οι Υπολογιστέ, ε, οι πληροφορικοί να χρησιμοποιηθούν περισσότερο. Και επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων. Και αυτό πρέπει να ε, το ε, διασφαλίσουμε και οι δημόσιες προμήθειε να είναι δίκαιε. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά. Και πρέπει να γίνει σαφέστερη η κατανομή και η οριοθέτηση αρμοδιοτήτων για να μην γίνονται επικαλύψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόσπισιλ είναι ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση. Μιλούμε για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θεωρώ ότι η ενιαία αγορά ήταν από τα βασικότερα επιτέγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και αν 28 χώρες καταφέρουν να συνεργαστούν, αυτό είναι καταπληκτικό. Και ακόμη και αν δεν είναι υπέρ μια πιο φεντεραλιστική Ευρώπη, θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα μεγάλα πλεονεκτήματα και τι ευκαιρίε που δημιουργεί η ενιαία αγορά για του πολίτε και τι επιχειρήσει. Ελπίζω και στο μέλλον να άρουμε τα εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία τη ενιαία αγορά και να ενισχύσουμε ίσω και κάποιε πτυχέ τη ενιαία ψηφιακή αγορά και να ρυθμίσουμε κάποια διασυνοριακά ζητήματα ιδιαίτερα των πωλήσεων ε, μέσω διαδικτύου. Και επίσης ε, να σταματήσει ο γεωγραφικός αποκλεισμός. Νομίζω ότι έτσι θα βελτιώσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ταυτόχρονα και την οικονομία μας. Ο κύριος Πόλτσακ, σας ευχαριστώ. Και εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Για τον απλούστατο λόγο ότι η ενιαία αγορά αποτελεί μια θεμελιώδη αξία και θεμελιώδες επίτευγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μάλιστα μετά από δεκαετίες προσπάθειες δίνει πολλά κίνητρα και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στους πολίτες αλλά και στις κυβερνήσεις για να προωθήσουν ε, περισσότερη ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστά αναφέρεται στην έκθεση η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, των επενδύσεων, αλλά και η πολιτική συνοχή αποτελεί ένα πόσπαστο τμήμα της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να μειωθούν οι ανισορροπίες και να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, καθώς και την καιροτομία. Όλα αυτά μας δίνουν μεγαλύτερη ενθάρρυνση για να συνεχίσουμε την ενιαγορά, αγορά. θα μας εξασφαλίσει ανάπτυξη οικονομική και απασχόληση. Περνάμε στο επόμενο θέμα, την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Τινησία. Κυρία Μορβά, ένα λεπτό. Λοιπόν, λοιπόν, άλλη μια λέξη για το λεξικό μου. Τι σημαίνει ελεύθερο εμπόριο. Ελεύθερο εμπόριο σημαίνει να μπορεί κανείς σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού να οθήσει τις ε, απολαβές προς τα κάτω για να μειωθούν και οι τιμές. Είτε πρόκειται για γεωργία, Βεβαίω για τη γεωργία σημαίνει πρέπει να καταστραφεί. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να καταστραφούν και οι εργαζόμενοι να μείνουν στην ψάθα. Ακόμη και ένα παιδί 4 ετών θα καταλάβαινε ότι όλα αυτά είναι εντελώ παράλογα. Γιατί δηλαδή πρέπει να εισαγάγουμε προϊόντα από μια χώρα που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Γιατί να μην αγοράσουμε προϊόντα που παράγονται πολύ πιο κοντά, χωρίς ε, παρασυτοκτόνα και άλλα τέτοια δηλητήρια. Θα ήταν πολύ καλύτερα να αγοράζουμε στην περιφέρειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαμίκης. Σας ευχαριστώ. Ιστορικά, η Ευρώπη και την Ισία ε, είχαν πάντα πολύ στενές σχέσεις τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις μας έγιναν ακόμη πιο στενές. Ξέρετε ότι υπήρξε αλλαγή καθεστώτος στην Τινησία και για την Τινησία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος, ιδιαίτερα για την διάθεση των γεωργικών της προϊόντων και κάθε χρόνο αυξάνεται αυτή η συνεργασία. Άρα πρέπει να κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα με βάση το πρόγραμμα για το ελεύθερο εμπόριο και λαμβάνοντας υπόψη αυτά που συνέβησαν στις 17 Μαρτίου όποτε, όποτε, όποτε και συνεδρίασε το Συμβούλιο Σύνδεσης Ένωσης στην Ισίας όπου συμφωνήθηκε όπως είπα ένα πρόγραμμα δράσης κάνουμε λοιπόν προσπάθειες να βοηθήσουμε περισσότερο την ε, Μεσόγειο ελπίζω να επιτύχει η συνεργασία μας ευχαριστώ πολύ παρακαλώ εσείς τώρα Ευχαριστώ, λέει ο Σκέλη, για μια ακόμη φορά. Υπερψήφισα με την ομάδα μου αυτές τις προτάσεις. Υποστηρίχθηκε η έκθεση από μεγάλη πλειοψηφία. 4,73 με 123 ήταν η διαφορά και τελικά υπήρξαν τέτοιες συμφωνίες με πολλές χώρες, παρόμοιες τέτοιες συμφωνίες, τις οποίες ψηφίσαμε και είναι σωστό να έχουμε και μια ανάλογη συμφωνία με την, την Ισία. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο επίμαχη αυτή η συμφωνία όπως άλλες, όπως είναι η TTIP, για την οποία υπήρξαν πολλές αντιρρήσεις και διαφωνίες και θα δούμε θα συμβεί. Με την Ισία είναι σωστό να προχωρήσουμε. Αλλά όπως είπε και η κυρία Μορβάη πρέπει να είμαστε προσεκτικοί δεν πρέπει να δημιουργήσουμε προβλήματα για τους Ευρωπαίους γεωργούς για να κάνουμε κάποια συμφωνία με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο δραστηριότητε του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και η κυρία Μορβά είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τους συναδέλφους να σκεφτείτε κάποιον ο οποίος περνάει δίπλα από μια λίμνη και βλέπει ε, πέντε να πνίγονται στη λίμνη. Και το άτομο αυτό αποφασίζει ότι πρέπει να σώσω έναν από τους πέντε. Το δικό μου το παιδί συγκεκριμένα. Είναι ηθική αυτή η απόφαση ή όχι. Από την άλλη μεριά δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Πέντε άτομα Ε, αν υπάρχουν πέντε άτομα που χρειάζονται φροντίδα και κάποιο φροντίσει του γονεί του από αυτού, τότε θεωρούμε ότι είναι ηθική αυτή η απόφαση. Εμεί στην Ουγγαρία και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε πιστεύουν ότι πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι είναι ναι με δύσκολη κατάσταση των προσφύγων, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε του δικού μα. Του δικού μα πολίτε συγκεκριμένα, του δικού μα ανθρώπου με τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι ηθική προσέγγιση. Και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κάνει αυτό. Ο κύριος Πόσπης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Μιας έκθεσης που παρουσιάζει διεξοδικά και περιγράφει τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητής, Ευρωπαίας Διαμεσολαβη... Διαμεσολαβήτριας εν Χαίρομαι που ενισχύονται αυτές οι δραστηριότητες και πολλαπλασιάζονται και είναι θετική αντίδραση και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στις συστάσεις. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί προς τι συστάσεις αν δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και δεν εφαρμόζονται. Χαίρομαι που 80% των συστάσεων ελήφθησαν υπόψη από τα θεσμικά όργανα και δόθηκε μια συνέχεια στις αιτιάσεις που υπευρέθησαν στην διαμεσολαβήτρια. Επίσης, ε, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να έχει δυνατότητα και μέσω του διαδικτύου να απευθύνεται άμεσα προς, τον, ε, προς την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Και ελπίζω αυτή η στενή επαφή με τους πολίτες να συνεχιστεί. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Το βασικό καθήκον του διαμεσολαβητή είναι να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής έχει όμως ευρύτερες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα το 2014 τα θέματα όπως θεμελιώδη δικαιώματα, το σύστημα των ε, λομπιστών και η διαφάνεια των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και η εγκύτητα των πολιτών προς την Ένωση ήταν τα σημαντικότερα θέματα. 20 με 30% των θεμάτων που τέθησαν στον διαμεσολαβητή είχαν να κάνουν με την ε, διαφάνεια. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι κάποια έγγραφα πρέπει να είναι διαβαθμισμένα και με περιορισμένη πρόσβαση. Αλλά όσον αφορά το TTIP δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν οι συζητήσεις να θεωρούνται διαβαθμισμένες. Αυτό δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο, Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ. Και πάλι χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να πω δύο λόγια για το θέμα της ε, Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, γιατί η Έμιλι Οράιλι είναι Ιρλανδέζα και έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο μέχρι στιγμής ε, ως διαμεσολαβήτρια. Μάλιστα, το 2014 είχαμε 2.163 αιτιάσεις που έτυχαν ανάλυσης και μάλιστα διεξοδικά από την κυρία Έμιλι Ράιλι και κατάφερε να διεκπαιρώσει πολλά θέματα και να βρει λύσεις για πολλά από αυτά τα παράπονα. Για μερικές περιπτώσεις μάλιστα ε, αποφάσισε να εκδώσει γνωμοδότηση και σε άλλες ε, να λάβει απόφαση. Χαίρομαι που είναι πενταετής πια ο χρονικός ορίζοντας της στρατηγικής για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και θα μπορέσει η κυρία Ράιλι να ξεκινήσει και κάποιες διαδικασίες αξιολόγησης. Εξαιρετικό το έργο της και τη συγχαίρω θερμά για, τις... για τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξήλθε στα καθήκοντά της. Και θα ήθελα να συγχαρώ και εσάς κυρία Πρόεδρε γιατί πραγματικά ε, προεδρεύσατε με άψογο τρόπο σήμερα. Συνεχίστε, συνεχίστε έτσι. Πάμε, προχωράμε, πάμε στο επόμενο σημείο το θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο κύριος Σούτη είναι που θα πάρει το λόγο αρχίσει η έκθεση του 2014 να συζητιέται το Φεβρουάριο του 2016. Διότι το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Δράγκη στην ουσία θα καταστρέψει το ευρώ με την πολιτική την οποία να ακολουθεί. Διότι κυκλοφορεί πολύ μεγάλη νομισματική μάζα, δεν μπορούμε να το πούμε αλλιώς αυτό, ως ε, τύπομα αλόγιστο χρήματος. Και όπως ξέρετε το επιτόκιο είναι μηδενικό. Αυτή η φλιβερή πολιτική του, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ε, το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν παίρνουν οι σωστοί άνθρωποι τις αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμη υποφέρουμε μετά από όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση. Έχουν υπάρξει εξελίξεις ε, που δυσχεραίνουν την οικονομική κατάσταση της Ένωσης. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν βοηθάει και υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Για παράδειγμα, η χρηματοδοτική πολιτική έναντι κάποιων κρατών μελών πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας αλλά δυστυχώς ε, φοβάμαι πως η περίοδος των παχαίων αγελάδων ε, ε, δεν θα συνεχιστεί στη Λετωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε στο νέο σημείο. Έναρξη διαπραγματεύσεων η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Μορβάη. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπερψήφισα για αυτήν την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Κάθε Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου είναι άλλη μία απόδειξη του τρόπου λειτουργίας ε, που ακολουθούμε ο τρόπος λειτουργίας μας θεωρείται ότι το χρήμα είναι τα πάντα. Δηλαδή όλοι θέτουν ως ερώτημα τι μπορώ να κάνω για να έχω περισσότερα κέρδη. Δεν έχουμε τον άνθρωπο στο κέντρο της προσέγγισής μας. Δεν ε, λειτουργούμε με βάση τι είναι καλό για το σύνολο, την, ε, το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Και όσοι έχουν τέτοια προσέγγιση πολύ συχνά είναι απεγνωσμένοι γιατί τόσο λίγες από τις συζητήσεις ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Εδώ έχουμε μείνει 5-6 άτομα. Σε ποιον μιλάμε σε αυτή την Ολομέλεια. Είναι πολύ λυπηρή η κατάσταση. Ο συνάδελφος είπε πρέπει να σκεφτούμε αυτά που λέμε εδώ πέρα. Τι λέω εγώ εδώ πέρα μέσα. Μιλάμε για ελεύθερο εμπόριο. Και το θεωρούμε κάτι το θετικό. Ακόμη και στο σχολείο μαθαίνουμε ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι κάτι το πολύ καλό. Αυτά μας λένε στο σχολείο. Θα πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση, πιστεύω. Και να αλλάξουμε την κατάσταση. Δεν πρέπει το χρήμα να είναι στο κέντρο της προσέγγισής μας, αλλά ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γεωγραφικά η Αυστραλία και η Νέα είναι πολύ μακριά βέβαια. Ωστόσο, από την αρχή του 20ου αιώνα έχουμε πολύ στενές σχέσεις με αυτές τις ε, περιοχές. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ανήκουν στο δυτικό κόσμο ε, και προσπαθούν να ε, διαφοροποιήσουν τις εμπορικές τους σχέσεις να αλλάξουν τις διοικητικές δομές της οικονομίας τους. Όλα αυτά δείχνουν ότι μπορούμε να τις προσεγγίσουμε και αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ιδιαίτερα εφόσον ε, τίθενται και θέματα φορολογικής, ε, συγγνώμη, νομοθετικής προσέγγισης. Άρα... Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε συμφωνήσει ελευθερία εμπορίο με δημοκρατία. Το Ηνωμένο Βασίλειο πλησιάζει όμω το δημοψήφισμα για να παραμείνει μέρο τη Ευρωπαϊκή συμφωνίε με χώρε κοινοπολιτή όπω ή όχι. Και συμφωνίε με χώρε κοινοπολιτή όπω η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι ιδιαίτερα πρόσδεκτε για πολλού από του ευρωσκεπτικιστέ συναδέλφου που στηρίζουν να χωρίσουμε μία από από, τις, από τα θετικά στοιχεία είναι ότι θα αυξήσουμε το εμπόριο με την κοινοπολιτεία με τη σφαίρα αγγλικής υπορροής. Η, η συμφωνία με τον Καναδά έχει ολοκληρωθεί και κινούμεθα προς τη διαδικασία κύρωσης. Οι διαπραγματεύσεις για το TIP συνεχίζονται και εδώ βρισκόμαστε τώρα να μιλούμε για συμφωνίες με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία να μην αναφέρουμε τον συνεχή ενθουσιασμό που υπάρχει για παρόμοια συμφωνία με την Ινδία δεν θα, δε θα εμποδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο να εμπορεύεται με την κοινοπολιτεία και άλλε χώρε. Η πρόθεση για συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω με άλλε χώρε θα κάνει το να είναι κανεί μέσω Ευρωπαϊκή Ενώσεω πολύ πιο υποφελή από ότι με μονομέ συμφωνίε του Ηνωμένου Βασιλείου με άλλε χώρε. Στη συμφωνία ΣΥΤΑ είδα ότι οι Καναδοί έκαναν παραχωρήσει που δεν υπάρχουν στι συμφωνίε ναύτα με τη ΣΥΠΑ. Και έχω την πεποίθηση ότι οι συμφωνίε με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα είναι εξίσου φιλόδοξε και επωφελεί για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα προχωράμε και πάμε στο θέμα των ζώων συντοφιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πρώτος που έχει το λόγο είναι ο κύριος Ντεμές Μάκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα ζώα συντροφιάς κάνουν τους, τα παιδικά τους όλο και πιο ε, χαρούμενους αλλά δυστυχώς τα ζώα είναι και αντικείμενο λαθρεμπορίου και αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες και θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να υπάρξει καταχώρηση και ταυτοποίηση των ζώων αυτών και είναι ένα κομμάτι του αναγκαίου μέσου που πρέπει να υπάρχει. Ανοίγει το δρόμο ε, όσον αφορά την καταχώρηση των σκύλων και των ε, ε, γατιών αυτό βοηθάει αν χαθούν τα ζώα να ξαναβρεθούν και να παρεμποδίσουμε το παράνομο εμπόριο που δεν σταματάει στα σύνορα. Γι' αυτό και το κόμμα μου υποστηρίζει περισσότερο μια ευρωπαϊκή δράση. Εάν έχουμε ε, καταχώρηση των κατοικιδίων ζώων με διαφορετικά μέτρα από χώρα σε χώρα είναι προβληματικό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το παράνομο εμπόριο και αυτό είναι υπέρ των ε, ζώων. Ο κύριος Πόσπης, ελέγχεται το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτή την πρόταση ψηφίσματος και χαίρομαι που υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ενιαίο μητρό ε, σκύλων και γάτων στην Ευρώπη. Θα καταπολεμήσουμε έτσι το λαθρεμπόριο των ζώων και τα βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται τα ζώα. δεν προσθέτουμε κάτι στην γραφειοκρατία, απλώς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα ζώα τα ζώα τα οποία κυρίως στην κεντρική Ευρώπη είναι αντικείμενο ε, λάθρεμπορίου, ε, γίνεται παράνομη αναπαραγωγή σε παράνομα κέντρα και μετάνουν στη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες άτυχα ζώα που ζουν σε φρικτές ε, συνθήκες. Εκεί γεννιούνται και μετά μεταφέρονται και παράνομα στη Δυτική Ευρώπη. Αν υπάρχει μητρό των ζώων, το λαθρεμπόριο των ζώων ε, θα υπόκει, μάλλον το εμπόριο των ζώων αυτών θα υπόκειται σε σαφείς κανόνες και η αντιμετώπιση των ζώων θα είναι καλύτερη. Θα τα θεωρούμε, θα αντιμετωπίζουμε σαν ζωντανά όντα και όχι σαν εμπορεύματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαμίκινς. Τα ζώα συντροφίας είναι τμήμα της καθημερινής μας ζωής. Είναι οι φίλοι μας. Είναι η βοηθή μας. Για ορισμένους ε, οι ανθρώπους ε, που είναι ίσως οι μόνοι φίλοι τους πολλοί δεν έχουν μόνο σκύλους και γάτες, αλλά έχουν χάμστερ, ε, ειδικά χειρίδια, ορισμένοι έχουν και κροκόδιλους και φίδια. Πρέπει λοιπόν ε, όμως κυρίως να επικεντρωθούμε στα πιο συνηθισμένα που είναι οι σκύλοι και οι γάτες. Επιτέλους εδώ και πολύ καιρό θα έπρεπε να υπάρξει τυποποίηση του συστήματος ε, καταγραφής σε όλα τα κράτη-μέλη, να υπάρχουν μητρώα δηλαδή. Αυτό θα βοηθήσει και την μεταφορά των ζών αλλά θα καταπολεμήσουμε με αυτόν τον τρόπο και το λαθρεμπόριο ζώων. Γιατί έχουμε τέτοιο πρόβλημα στην Ένωση και είναι πολύ σημαντικό. Περνάμε στο τελευταίο θέμα σήμερα, την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη. Η κυρία Μορβά είναι η πρώτη ομιλήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω επικρίνει τις αποφάσεις μας, τις αποφάσεις μας για πολλά θέματα. Να πω και κάτι θετικό. Θεωρώ, με βάση αυτά που άκουσα, ότι έχουμε αλλάξει τρόπο προσέγγισης. Και αυτό φαίνεται στην ε, έκθεση για την Ιεμένη. Ε, η Ένωση θεωρεί ότι για συγκεκριμένους λόγους σε μια χώρα στον τρίτο κόσμο έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν ε, προσφυγικές ροές από αυτή τη χώρα και εμείς θα πρέπει να δεχθούμε αυτές τις ροές. Εάν μια χώρα όπως η Ουγγαρία δεν δέχεται τέτοιες ε, προσφυγικές ροές, τότε η χώρα αυτή είναι αντικείμενο επικρίσεων από τους εταίρους της. Στην έκθεση για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη ωστόσο, στην Ιωμένη ωστόσο επιτέλους ε, ε ονομάζουμε τα πραγματικά αίτια. Και εδώ είναι σαφές ότι η στρατιωτική παρέμβαση διαφόρων οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, την καταστροφική στην Ιεμένη. Επιτέλους ε, επικρίνουμε την Σαουδική Αραβία και το εμπόριο όπλων που κάνουν πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτός ο τρόπος να αναφέρουμε και να αντιμετωπίσουμε τα αίτια και όχι να επικρίνουμε αυτούς που δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν να υποδεχτούν πρόσφυγες. Μα Μίκινς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι για δεκαετίες η Εμένη ήταν μία από τις φτωχότερες ε, χώρες του κόσμου. Η επανάσταση πριν από πέντε χρόνια όχι μόνο δεν βελτίωσε, αλλά αντίθετα επιδίνωσε την κατάσταση. Και οι τελευταίες παρεμβάσεις ε, της Σαουδικής Αραβίας και η στήριξη του Ιράν για τους ε, Χούτι επιδίνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους κατοίκους αυτής της χώρας δεν ε, είναι σαφής η εξέλιξη της, ε, των σειράξεων. Είναι λοιπόν τραγική η ανθρωπιστική κατάσταση. Αν θέλουμε να μην υπάρξει ανθρωπιστική καταστροφή, πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει ένα ουσιαστικό εμπάργο. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο προς έγκριση στις αρχές της επόμενης ε, συνεδριάσεως και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα προωθήσω τα εθετηθέντα ψηφίσματα της σημερινής συνεδριάσεως στους ε, φορείς και τους ανθρώπους